Hello, good morning. Please be welcome. Be welcome. Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω. Ας ξεκινήσουμε με τις εργασίες μας με ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω στις ανακοινώσεις ότι είχαμε ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο για την εκτελεστική απόφαση ως προς την ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών στοιχείων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η προθεσμία τροπολογιών είναι για σήμερα στις 9.30. Έχουμε λάβει δύο τροπολογίες Άρα, ως εισηγητής, θεωρώ ότι επειδή είχαμε ανταλλαγή απόψε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και στην ουσία δεν είχαμε και αυτά αποτελέσματα ή επαρκής διασαφηνήσεις και δεν μπορούσε να μας πει το Συμβούλιο πότε, πότε θα αρχίσει η αυτόματη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών στοιχείων με το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε πόσα κράτη-μέλη θα ευεργετηθούν από αυτή την ανταλλαγή απόψεων το 2020 κατά την ε, μεταβατική περίοδο και δεν μας μίλησε και για ρήτρες ασφαλείας που θα ισχύσουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ως προς την ανταλλαγή δεδομένων με το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης ασφάλειας. Θα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες από το Συμβούλιο, γι' αυτό αναβάλω τη σημερινή ψηφοφορία, όπως συμφωνήσαμε με τους Σκιώδης, μέχρι ότου λάβουμε περισσότερες πληροφορίες από το Συμβούλιο. Προχωράμε λοιπόν με το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Είναι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών. Ο κύριος Σαρσαλέχος είναι ο εισηγητής. Θα αρχίσουμε όμως με την ουσία της ε, ανταλλαγής απόψεων, γιατί πρόκειται για ένα μέσον που ε, οδηγεί στην ε, αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα του ποινικού δικαίου και δείχνει ότι υπάρχουν και κενά. Κενά στον τομέα του ποινικού και ιδιαίτερα σε σχέση με ορισμένα υποτιθέμενα προβλήματα ως προς τις συνθήκες φυλάκισης, τον ορισμό της ε, δικαστικής αρχής, τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την πρόσβαση σε συνήγορο και τις διαφορετικές έννοιες ως προς την ε, ανεξαρτησία των εισαγγελικών αρχών. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να σταθούμε σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση και μεταρρύθμιση του τομέα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Σύλληψη. Σήμερα έχουμε τρεις ε, εμπειρογνώμονες που θα μας μιλήσουν για το θέμα, τον κύριο Βάουτερ Βαν Μπαλεγόη, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής της Μονάδας Ευρωπαϊκής Προσθέμενης Αξίας, την κυρία Ιβάνα Κίντλ Κρίστο, από την ε, Πολιτική Υπηρεσία και την Γενική Διεύθυνση ε, Δικαιοσύνης και τον κύριο Φρανσκίσ, Φρανθίσκο Χιμένες Βιγιαρέχο, που είναι μέλος της ε, Eurojust. Μετά θα έχουμε συζήτηση και το γύρο έρωτα αποκρίσεων από τον εισηγητή και του Σκιώδης. Αλλά πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ακούσουμε από τον εισηγητή μας, από τον κύριο Σαρσαλέχος, ο οποίος έχει και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους τους παριστάμενους, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον εκπρόσωπο της Eurojust και τον ε, εκπρόσωπο των ε, μελετών του Ευρωκοινοβουλίου που έκανε μια πολύ ουσιαστική εργασία και η οποία και θα συνεχιστεί. Ήδη έγινε μια πρώτη συνάντηση με τους Σκιώδη σε σχέση με την έκθεση αυτή, με ανταλλαγή απόψεων και φυσικά δεν υπάρχουν πάντα συγκλίνουσες ε, θέσεις, ε, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία, αλλά υπάρχει ένα κοινό έδαφος για τους ε, τομείς όπου μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις. Έχουν περάσει 18 ε, χρόνια από τότε που τέθηκε αυτό το πλαίσιο και 16 χρόνια από τότε που ετέθησε σε ισχύ. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και παράλληλα μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε επί της ουσίας για δύο δεκαετίες σχεδόν η εισαγωγή αυτού του μέσου δικαστικής ε, συνεργασίας που βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση, μια εγκάρσια αρχή, αλλά ε, δεν μπορεί να υπάρχει αναγνώριση αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός υπό την έννοια ότι η εμπιστοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού του οικοδομήματος μέσα στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας για να φτάσουμε σε έναν αποτελεσματικό χώρο ελευθεριών. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις στην απόφαση πλαίσιο. Δεν ε, υπάρχουν ε, διαρθρωτικά σφάλματα δηλαδή σε αυτό το μέσο, αλλά ως προς την εφαρμογή του ε, θεωρώ ότι υπάρχουν ελλείψεις, όπως δείχνει και αυτή η έκθεση. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε μερικές. Μιλάμε για ζητήματα όπως την ερμηνεία της εφαρμογής των, ε, της ενδεχόμενης απόρριψης ενός εντάλματος σύλληψης και επίσης θέματα αμοιβαίας εμπιστοσύνης των ε, δικαστικών αρχών και η διαφορετικότητα του ποινικού δικαίου και της ερμηνείας του μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και ο κατάλογος αδικοπραξιών για να μην υπάρχει ε, διπλή ε, διπλέ, για να μην υπάρχουν διπλές καταδίκες και γι' αυτό ακριβώς θα μας απασχολήσει το ε, θέμα μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των δικαστικών αρχών για ένα πιο ευέλικτο μέσο το οποίο να μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίπτωση όταν ορίζουμε αυτή τη συνεργασία. Το ευρωπαϊκό ένταλμα λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα των, του ποινικού στα κράτη-μέλη και της εσωτερικής ένομης τάξης, αλλά ε, η απόφαση πλαίσιο μας επέτρεψε να λειτουργήσουμε με βάση τη διαφορετικότητα του ποινικού δικαίου στα κράτη-μέλη. Έχουμε ευρύτατη πείρα ως προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος και θα πρέπει να δούμε ποιες ε, είναι οι νέες προκλήσεις μες στα πλαίσια της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και ως προς το, την ψηφιακή μορφή του εγκλήματος και θα πρέπει να δούμε και την εξέλιξη και των νομοθεσιών και των ορισμών νέων εγκλημάτων και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη σημαντική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που βοήθησε αποφασιστικά στη, ως προς την ε, πρακτική εφαρμογή του εντάλματος και όλα αυτά υπό την προοπτική των θυμάτων, τα δικαιώματα των οποίων δεν μπορούμε να αγνοήσουμε λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές φορές μπροστά στις νέες μορφές εγκληματικότητας βλέπουμε ότι δεν ικανοποιούνται τα θύματα και δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το δικαστικό μέσο να υπηρετεί τα θύματα πρωτίστως. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο σκέψης μας και μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, γι' αυτό θα συνεργαστούμε για την έκθεση αυτή και θα υποβάλω την έκθεση τον Απρίλιο. Ευχαριστώ κύριε Θαρσταλέχος για την παρουσίασή σας. Περνάμε αμέσως στη συνέχεια για να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο με τη σειρά ε, στα μέλη του πάνελ εδώ στους ομιλητές μας. Ακούσουμε πρώτα για 12 λεπτά το δόκτωρα Βάουτερ Βαν Μπάλεχόη, πολιτικό αναλυτή στη Μονάδα Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υπό την ιδιότητά μου αυτή θα ε, μιλήσω για την ε, ε, μονάδα ανάλυσης εκ των υστέρων. Καλά, αυτό είναι λεπτομέρεια. Ε, σας ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη αυτή η στιγμή σήμερα για μένα γιατί πριν από 17 χρόνια όταν άρχισα την ε, ακαδημαϊκή μου καριέρα στη Χάγη, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο, μας προσέγγισε ένας Ολλανδός δικαστής και μας είπε ότι θέλω να γράψω κάτι για αυτό το περίεργο εργαλείο που βγάζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, ε, εγώ δεν ήξερα ότι ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δικαστική συνεργασία. Νόμιζα ότι ασχολείται μόνο με ε, τις πτυνοτροφές. Ε, εν πάση περιπτώσει, έκανα και το διδακτορικό μου για την αμοιβαία αναγνώριση και τελικά αυτό με οδήγησε να μιλώ σήμερα στην Επιτροπή σας ως μέλος της Μονάδας Ερευνών. So, um, can we go to the first slide? Ε, μπορούμε να περάσουμε ε, στην πρώτη διαφάνεια. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω σήμερα την ανάλυση αυτή σε ε, βάθος που συνέταξα μαζί με τη συνάδελφο Ιβάνα Κίντλ, εδώ παρακαθήμενη. Όπως είπε ήδη ο, ο είναι μια διαδικασία που περνά από διάφορε φάσει. Αυτή είναι μια πρώτη ανάλυση με κάποια πρώτα ευρήματα. Παρακαλώ, ω τέτοια να την εκλάβετε. Ε, τον Απρίλιο, μαζί με την τελική έκθεση, θα έχουμε πιο ε, βαθιά μελέτη για ε, οτιδήποτε έχει να κάνει με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψης και ήδη από τώρα μπορώ να σα ανακοινώσω ότι είναι αυτά πολλά. Ε, λοιπόν, παρακαλώ να παραμείνουμε σε αυτή τη διαφάνεια, στην προηγούμενη δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, Φυσικά, τα ε, ευρωπαϊκά κράτη εδώ και δεκαετίες, ε, μάλιστα αιώνες, εκδίδουν ε, το ένα στο άλλο πολίτες με βάση τις διεθνείς συμβάσεις. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω να κοιτάξετε την αριστερή στήλη, την κόκκινη, που δείχνει κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις εκδόσεις όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτον, ήταν πολύ αργές αυτές οι διαδικασίες. Καμιά φορά χρειαζόταν και ένα ολόκληρο έτος για να εκδοθεί κάποιος από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο. Ε, δεύτερο πρόβλημα ήταν ε, πάρα πολύ βαριές οι διαδικασίες αυτές με συμμετοχή πολλών προσώπων έτσι ώστε να επιτευχθεί η έκδοση του ενδιαφερομένου. Τρίτο, πολύ σημαντικό, ε, αρχή όλων αυτών ήταν η αρχή της εθνικής κυριαρχίας. Κυρίαρχα κράτη αποφάσιζαν μεταξύ τους αν μπορούσε κάποιο να εκδοθεί ή όχι. Και υπήρχαν φυσικά ε, και κάποιες εξαιρέσεις ε, με βάση την ηθαγένεια. Δηλαδή ότι εμείς δεν εκδίδουμε πολίτες που έχουν την ηθαγένεια του κράτους μας. Κάτι το οποίο και πάλι είναι επίκαιρο στις συζητήσεις που γίνονται για το Brexit. Η, ε, η διπλή δίωξη, το ξανακούσαμε και προηγουμένως. Δηλαδή θα πρέπει να συγκρίνουμε ε, με το δικό μας ποινικό σύστημα εάν αυτές οι πράξεις είναι αξιόπινες και στη δική μας χώρα πριν αποφασίσουμε εάν και κατά πόσο θα εκδώσουμε κάποιον. Ε, το διπλό αξιόπινο λοιπόν. Ε, Τι έχουμε δει όμως από τη συνθήκη του Άμστερνταμ και μετά. Υπάρχει φιλοδοξία οικοδόμηση ενό χώρου ασφάλειας, ελευθερία και δικαιοσύνης. Έχουμε ένα ενιαίο νομικό χώρο πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξού και η αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης. Τι σημαίνει αυτό καταρχήν, ότι θα πρέπει να εκτελεί κανεί ένα ένταλμα που έχει εκδώσει άλλο κράτο μέλο. Καταρχήν, θα επανέλθω στη συνέχεια σε αυτό. Τι έχει γίνει λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν, ε, όπου χρειαζόταν περίπου ένα χρόνο. Τώρα έχουμε φτάσει στι 40 ημέρε ε, ε, όταν διαφωνεί ο ενδιαφερόμενος και γίνεται ακρόαση πριν την παράδοσή του. Υπάρχει ένα στάνταρ έντυπο που έχουμε για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο και σας δείχνω, και οδήγησε σε πάρα πολύ μεγάλη απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης που ονομάζονται διαδικασίες παράδοσης γιατί έχουμε μια κοινή ε, πλέον ε, δικαστική συνεργασία και έναν ενιαίο ε, νομικό χώρο. Και φυσικά έχουμε ξεφύγει από την πολιτική λήψη απόφασης προς τη δικαστική λήψη απόφασης. Ανεξάρτητες δικαστικές αρχές συνεργάζονται και αποφασίζουν εάν κάποιος μπορεί να παραδοθεί ή όχι. Παρόλα αυτά, ε, παραμένουν οι προκλήσεις. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά με την αμοιβαία αναγνώριση κυρίως, αλλά και την έννοια των δικαστικών αρχών. Θα ε, επανέλθω στη συνέχεια στα προβλήματα. Ε, πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Ε, θα ασχοληθώ με τρεις βασικές προκλήσεις ή προβλήματα. Υπάρχει αυτή η μικρή έκδοση, υπάρχουν πολλές ακόμα, αλλά έχουμε 12 λεπτά στη διάθεσή μας. Λοιπόν, ε, ποιε είναι οι ανεξάρτητες ε, δικαστικές αρχές. Δεύτερον, σχέση ε, ανάμεσα στην αμοιβαία αναγνώριση, την εναρμόνιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και της ποινική δικονομία. Και το τρίτο, η αμοιβαία αναγνώριση και σχέση με την συμμόρφωση προ τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε ακούσει ήδη ότι πριν από 18 χρόνια ε, έγινε το προσχέδιο κειμένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Ωστόσο, μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσπαθούσε να ορίσει τι εστί ανεξάρτητη δικαστική αρχή, δηλαδή ποιος μπορεί να εκδώσει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πολύ ε, σύντομα. Ας πούμε, ένας Γάλλος, ένας Σουηδός, ένας Γερμανός, ένας Βέλγος εισαγγελέας είναι αρκετά ανεξάρτητος. Όλες αυτές οι ερωτήσεις έχουν φτάσει ως προδικαστικά ερωτήματα στο δικαστήριο μέχρι πολύ πρόσφατα. Και ήδη το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι τα αστυνομικά όργανα και τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας σίγουρα δεν θεωρούνται ε, ε, ε, εκδίδουσες μάλλον αρχές δικαστικές ανεξάρτητες και έχουν ορίσει κάποια κριτήρια. Είμαι σίγουρος ότι ο συνάδελφος της Eurojust θα επεκταθεί στη συνέχεια σε αυτό και θα σταματήσω εγώ εδώ γι' αυτό. Ε, το κοινοβούλιο σας επίσης ε, έχει κάποιες ανησυχίες ε, σε σχέση με την αναλογικότητα, δηλαδή του αριθμού των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί. Αυτό έχει δύο πόλους. Από τη μια όλα τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, ακόμα και αν είναι θεμητό να σταλούν, ε, είναι αναλογικά. Και δεν θα σας ε, κοροϊδεύω σας έλεγα ότι ένας κλεφτοκοτάς, ας πούμε, ή κάποιος που δεν πληρώνει το ξενοδοχείο του, στο παρελθόν ε, ε διώκεται με ε, ένταλμα σύλληψη ευρωπαϊκό. Αυτό μπορεί να θεωρείται απώλεια χρόνου και ενέργεια, αν σκεφτεί κανεί ότι η διαδικασία αυτή κοστίζει 25.000 ευρώ. Επίσης, τώρα ερχόμαστε στα ποινικά και ποινική δικονομία και τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πότε έχει ολοκληρωθεί η δίωξη ποινική ε, και μπορεί κάποιο να παραδοθεί. Ε, είναι τελείω διαφορετική η κατάσταση από χώρα σε χώρα και Γι' αυτό, de facto, καλούν κάποιου ακρόαση αντί να του στέλνουν στην ακροματική διαδικασία, σε ένα δικαστήριο. Ε, το Κοινοβούλιο κάποια στιγμή έχει κάνει ε, μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλία και ζήτησε να ε, μεταρρυθμιστεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε με ένα εγχειρίδιο λέγοντας ότι βεβαίως μπορούμε να έχουμε κάποια κριτήρια που να εφαρμόζονται πριν αποφασίσει η εκδίδουσα αρχή εάν πρέπει να εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψη ευρωπαϊκό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να πούμε ότι ήταν ε, ικανοποιητική ε, αυτή η ε, διαδικασία. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Um, Επίσης, οι ύποπτοι όταν παραδίδονται θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα δικαστούν με τρόπο ε, αμερόληπτο και ανεξάρτητο. Ένα Ιρλανδικό δικαστήριο επίσης έκανε ένα ερώτημα ε, σε σχέση με μια παράδοση στην Πολωνία και ρώτησε λοιπόν το δικαστήριο έχω ε, κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε. Ακόμα και αν η λόγω χώρα είναι υπό τη διαδικασία του άρθρου 7.1, ε, θα πρέπει κατά περίπτωση να ε, ελεγχθεί εάν θα είναι αμερόληπτη και ανεξάρτητη δίκη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού συνεννοήθηκαν οι δικαστικές αρχές μεταξύ τους, διαπιστώθηκε ότι έχει αρκετές εγγύησεις ο Ιρλανδός δικαστής για να πει ότι κοιτάξτε, το συγκεκριμένο δικαστήριο θα είναι και ανεξάρτητο και αμερόληπτο, οπότε παραδόθηκε στην Πολωνία ο ενδιαφερόμενος. Και πάλι αυτό είναι μια πολύ πρόσφατη απόφαση για ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Και ποιο είναι το επίκαιρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φέρει ε, την πρώτη έκθεση, ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου. Και το Κοινοβούλιο ζήτησε έναν ευρύτερο μηχανισμό ε, για την, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ έχουμε το ακαθόδες θέμα του διπλού αξιόπινου αυτό έχει να κάνει ε, με ε, την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Ε, βλέπουμε την αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης και δεξιά βλέπουμε τι έκανε η περίφημη απόφαση. Δεν εφάρμοσε πλήρως αυτή την έννοια. 32 κατηγορίες αξιόπινων πράξεων το έπραξε που θεωρούνται αρκετά σοβαρές από την ε, νομολογία του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έτσι ώστε να ε, δοθεί εντολή, να παραδοθεί ο διαφερόμενος. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως η εναρμόνιση της αξιόπινης πράξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ε, Είναι πολύ καλή η απόφαση πλαίσιο, καλή ως παράδειγμα, για το οργανωμένο έγκλημα. Τι είναι το οργανωμένο έγκλημα? Σε ένα εναρμονισμένο σύστημα. Το εναρμονισμένο σύστημα δεν είναι το άθροισμα των ε, εθνικών διατάξεων. Η εξαίρεση είναι το άρθρο 4.1 ε, της ε, απόφασης πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχει οδηγήσει σε πολλή συζήτηση για την εντολή που δίνει εκδούς αρχή να εξετάσει Πώς ορίζεται αυτή η αξιόπινη πράξη στη χώρα που εκδίδει το ένταλμα και πώς ορίζεται στη χώρα που ε, εκτελεί το ένταλμα σύλληψη. Αυτό όμως είναι σύμβατο με την αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης, οπότε θα πρέπει να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, να αποφανθεί ε, για το βαθμό ομοιότητας που έχουν αυτά τα δύο στις δύο χώρες. Η συζήτηση σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Ε, Προχωρούμε στην επόμενη διαφάνεια. Δεν ξέρω, μετράτε. Έχουμε πολλά ε, νομικά εργαλεία, μια τουζίνα και παραπάνω αρχίζοντας από ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συνεργασίας. Έρχομαι τώρα στην συνεργασία στην ποινική δικαιοσύνη. Τελειώνω, τελειώνω. Ε, βλέπουμε ότι ε, έχουν εγκριθεί πολλά μέσα και εργαλεία και θα επιταχύνω λίγο τώρα ε, σε ό,τι αφορά τη διερμηνία και τη μετάφραση, την ενημέρωση στις ποινικέ διαδικασίες, πρόσβαση σε συνήγορο, ανήλικη και νομική αρρωγή. Όπως βλέπουμε, η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία ε, και η ε, εφαρμογή ακόμα εχολένουν. Και πάω στην τελική μου διαφάνεια και επανέρχομαι στη συζήτηση που είχαμε για τα ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια και τώρα μιλούμε για τις συνθήκες κράτησης. Η αμοιβαία αναγνώριση ε, απαιτεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαία εμπιστοσύνη σημαίνει ότι τα διεθνή πρότυπα κράτησης στηρούνται και εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη-μέλη. Άρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, έχει εκδώσει κάποιες αποφάσεις που δεν κρατούν τα κράτη, ε, τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κράτησης και το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απαντήσει. Αυτό ακριβώς έκανε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την υπόθεση αραιώση και ε, στη συνέχεια εξελίχθηκε. Και εδώ έχουμε φτάσει στο να συζητάμε πόσα τετραγωνικά μέτρα αναλογούν ανακρατούμενο σε ένα κελί όπου συστεγάζονται πολύ ε, κρατούμενοι. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ. Βλέπω πως προσπαθείτε να με βοηθήσετε για να διαχειριστούμε και τη χρονική διάρκεια αυτής της ακρόασης για το ευρωπαϊκό ένταλμα. Και με τον τρόπο αυτό και όλοι οι πανελίστες θα εκφραστούν και τα μέλη θα μπορέσουν να πάρουν μέλος στη συζήτηση. Περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο ε, μέλος αυτού του πάνελ από τη Γενική Διεύθυνση ε, Justice. Σας δίνω λοιπόν το λόγο σας ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Αγγιλάρ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ για ένα εργαλείο το οποίο είναι σημαντικό και είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Πολύ συχνά το αναφέρουμε ως το εμβληματικό εργαλείο στην δικαστική ε, συνεργασία για ποινικά θέματα. Ο, ο, ο μιλητής δίπλα μου αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν από την ε, συνδρομή και την εκτέλεση και διάφορα θέματα προκύπτουν από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου αλλά και από το ψήφισμα του 17 για τις συνθήκες στις φυλακές. Να σας πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει σε βάθος τα θέματα αυτά και θα ήθελα να υπογραμμίσω πως τα προβλήματα που έχουμε με την εκτέλεση του, συντα... Ε, του εντάλματος ε, δεν είναι τόσα πολλά, είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο στα πλαίσια της δικαστικής συνδρομής και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα. 7.000 περίπου εκτελέστηκαν το 2005 και αυτός έχει φτάσει σε πάνω από 17.000 το 2018. 7.000 ε, εκτελέστηκαν, οπότε θα έλεγα πως 40% από τα εντάλματα που εκδόθηκαν εκτελέστηκαν. Θα πω λοιπόν κάτι παραπάνω για τα στατιστικά δεδομένα, γιατί θεωρώ πως μπορεί να προκαλέσουν κάποια σύγχυση γιατί μπορεί κανείς να θεωρήσει πως αν το 60% των ενταλμάτων είναι ανεκτελεστά, τότε ε, το εργαλείο δεν λειτουργεί. Δεν ισχύει αυτό. Καταρχήν, αρκετά συχνά εκδίδεται το ευρωπαϊκό ένταλμα, αλλά δεν μπορεί να εντοπιστεί ο κατονομαζόμενος ε, ε, άνθρωπος, γιατί έχει εξαφανιστεί. Δεύτερον, τα όσα έχουν εκτελεστεί μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ε, κάποια που έχουν εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά αλλά έχουν εκτελεστεί την επόμενη ή και δύο χρόνια μετά γιατί τότε ε, βρέθηκε το άτομο για να ε, συλληφθεί και πολλές φορές έχουμε και πολλαπλά εντάλματα στο ίδιο όνομα. Άρα λοιπόν, αν το άτομο έχει ήδη παραδοθεί ή συλληφθεί, ένας μεγάλος αριθμός απλώς δεν εκτελείται. Επίσης, υπάρχουν και λόγια απόρριψης που έχουν να κάνουν με το γεγονός πως το άτομο δεν βρέθηκε. Και πρέπει να σας πω πως είναι το άρθρο 4.6 που είναι ο βασικότερος λόγος απόρριψη που επιτρέπει ε, ε, υπηκόους και διαμένοντες να μην παραδίδονται και να μην εκδίδονται αρκεί ε, το κράτο μέλος να αναλάβει να εκτελέσει την ποινή το ίδιο. Άρα λοιπόν το ένταλμα θα απορριφθεί αλλά δεν σημαίνει αυτό πως θα οδηγηθούμε σε ατιμορρησία εκτελείται από το οικείο κράτος μέλος. Επίσης, έχουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτά χρησιμοποιούνται και τα επικαλείται και η Γερμανία τα τελευταία χρόνια και θα το ε, παρουσιάσω σε βάθος. Επίσης, καμιά φορά είναι δύσκολο να συγκρίνουμε από χρόνο σε χρόνο τα αριθμητικά στοιχεία. Γιατί, Γιατί δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να στείλουν τα δεδομένα αυτά, γίνεται σε εθελοντική βάση, οπότε κάποια κράτη-μέλη δεν στέλνουν στατιστικά κάθε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή εξετάζει τη δυνατότητα να ε, χρησιμοποιηθεί μία ε, πλατφόρμα ε, ψηφιακή η οποία αυτή τη χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική μαρτυρία και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για να συμπεριλάβει και το ευρωπαϊκό ένταλμα και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να λαμβάνουμε και καλύτερα και πιο συγκρίσιμα στοιχεία στο μέλλον. Έχει ήδη αναφερθεί και θα το πω πάλι, η νομολογία του ΔΕΚ έχει αυξηθεί ριζικά τα τελευταία πέντε χρόνια και ενώ είχαμε μόνο 15 υποθέσεις το 14 που πέρασαν από το ΔΕΚ, Τώρα έχουμε πάνω από 50 υποθέσεις στις αρχές του 2020. Δεν είναι πάντα εύκολο για τους ε, νομικούς ε, να παρακολουθούν την ε, νομολογία, αλλά επιτρέπει στο ΔΕΚ να ξεκαθαρίσει θέματα που έχουν να κάνουν με την ισορροπία μεταξύ της αμοιβαίας συνδρομής και του σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τώρα έχουμε και κάποια πιο προβληματικά θέματα, τα οποία έχουμε εντοπίσει και αυτό έχουν να κάνουν με το ένταλμα και μπορούμε να τα μοιράσουμε σε δύο κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα τα θέματα που προκύπτουν με την ατελή ή εσφαλμένη ε, εφαρμογή της απόφασης. Στην πρώτη αυτή κατηγορία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία μελέτη συμμόρφωσης ε, στις εθνικές νομοθεσίες και το πώς έχουν μεταγράψει το ευρωπαϊκό ε, ένταλμα το 18-19 και πάνω στα στοιχεία αυτής της μελέτης θα παρουσιάσουμε μια έκθεση ε, εφαρμογή, την οποία θα δημοσιεύσουμε ελπίζω πριν το καλοκαίρι φέτο. Η έκθεση αυτή μαζί με άλλες εκθέσεις ε, στα θέματα του ποινικού και ε, δικαίου και για σχετικά δικανικά θέματα θα είναι πολύ σύντομη, 15 σελίδες, δεν θα κατονομάζονται κράτη-μέλη και δεν θα είναι πολύ περιγραφική. Θα δώσει μια επισκόπηση των πιο προβληματικών θεμάτων ε, στην μεταγραφή της ε, εφαρμοστικής ε, απόφαση, της απόφασης αυτής, με θα είναι συμπληρωματική με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς θα μιλήσετε για τα πρακτικά κενά στην εφαρμογή του εντάλματος, ενώ η δική μας έχει να κάνει με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Να σας πω πως η πρώτη μας ανάλυση έδειξε πως τα θέματα μεταγραφής έχουν να κάνουν με τα συγκεκριμένα εξή θέματα. Πρώτον, λόγια απόρριψης, οι οποίοι εφαρμόζονται υποχρεωτικά, ενώ θα έπρεπε να αποτελούν εναλλακτική λύση. Δεύτερον, κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, προσθέσει ε, λόγους απόρριψης και κυρίως απαγόρευση παράδοσης υπηκόων αλλά και παρά, ε, ε, ε επίσης ε, ανθρώπινα δικαιώματα, αναλογικότητα και διάρκεια δικαστικής διαδικασίας. Να σας πω πως το διπλό αξιόπινο είναι εκτός πεδίου των εργαλείων και έχουμε πολλές φορές και ε, προβλήματα με τις υποχρεώσεις με τις που προκύπτουν από τις προθεσμίες που δίνονται για τις διάφορες φάσεις της δικαστικής διαδικασίας και κυρίως ε, της διαδικασίας εφέσεων. Και πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές και κάποια κομμάτια της νομοθεσίας δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά. Δεύτερη κατηγορία θεμάτων που προκύπτουν και έχουν κάνουν με την εσφαλμένη εφαρμογή του εργαλείου. Κάποια ε, αναφέρθηκαν από τον κύριο Μπαλιχόη, αλλά θα σας πω η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύει. Πρώτα απ' όλα, αναλογικότητα. Οι διαφορές που προκύπτουν με την αναλογικότητα και την αξιολόγηση αυτής εξηγούνται από τις επιλογές που κάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με την δίωξη και τις πολιτικές δίωξη. Κάποιοι έχουν κακολουθεί στην αρχή της νομιμότητας και την υποχρεωτική δίωξη ή την αυταπάγγελτη ε, δίωξη και οι άλλοι είναι η καθευκαιρίαν. Έτσι λοιπόν η πλειοψηφία των κρατών μελών έχουν ε, κάνει επιλογές και μηχανισμούς στα ε, ε, συστήματά τους έτσι ώστε να μην εκδίδονται τέτοια εντάλματα για, αδικήματα, για ίσον αδικήματα. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για να μειωθεί η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Έχουμε και κάποιες ενδείξεις από τα στατιστικά πως το πρόβλημα μειώνεται αυτή τη στιγμή 4.800 ε, εντάλματα έκδοσε το 2009 η Πολωνία και το 18 μόνο 2.300. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε μία μείωση ε, πάνω από 50%. Όταν όμως έχουμε βασικές ανησυχίες για την αναλογικότητα, τότε μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει και σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο. Δηλαδή, η δική μας συμβουλή στο εγχειρίδιο των αθεωρημένων του 17 λέει πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μία σειρά κριτηρίων πριν αποφασίσουν τι θα κάνουν με το ένταλμα και αν θα εκδώσουν ευρωπαϊκό ένταλμα. Επίσης, η, εκτελ εκτελούσες αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη πως χρειάζεται να επικοινωνήσουν με την ε, χώρα έκδοσης και βέβαια η χώρα έκδοσης θα πρέπει πριν παραδώσει το άτομο να έρθει σε επαφή με την χώρα έκδοσης του εντάλματος. Για τα θεαμιλιώδη δικαιώματα και όσα προκύπτουν εκεί αναφέρθηκε, έχουν, είναι ένα εργαλείο αμοιβαία αναγνώρισης, χρειάζεται αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών και ε, βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει φανεί πως η αμοιβαία εμπιστοσύνη έχει κάποιους περιορισμού αυτό που διαπιστώνουμε είναι πως υπάρχει μια αυξανόμενη τάση στα κράτη-μέλη στις διοριακές διώξεις να μην εμπιστεύονται το ένα το άλλο και κυρίως για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Ουγγαρία, ε, Ρουμανία έχουμε και πολλά παραδείγματα. Κάποια κράτη-μέλη, Γερμανία, Αυστρία, κάτω χώρες και Ιρλανδία είναι όλο και πιο διστακτικά να εκτελέσουν με αυτόματο τρόπο αποφάσεις ε, για ευαίσθητα ποινικά θέματα. Άλλα κρατημέλη, όπως για παράδειγμα η Γαλλία και η Ισπανία, ανισχούν ιδιαίτερα από το γεγονός πως η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης παραμερίζεται και με τον τρόπο αυτό μειώνεται η αποτελεσματική συνεργασία σε ποινικά θέματα. Ένας λόγος ο οποίος αναφέρθηκε πριν από αυτή τη μειωμένη εμπιστοσύνη και ένας από τους βασικούς λόγους και για τους οποίους είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε το κράτος δικαίου είναι οι ε, συνθήκες κράτησης ε, και οι υπεράριθμοι κρατούμενοι στις φυλακές των κρατών μελών. Αυτό ξεκαθαρίστηκε τώρα από το ΔΕΚ ε, στην απόφαση Αλαντιόζη, όπως επίσης και σε δύο ακόμα αποφάσεις και πρέπει να σας πω πως ε, πρέπει να δούμε τι συνέβη μετά από αυτές τις αποφώσεις του ΔΕΚ με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα. Καταρχήν, οι συνθήκες φυλάκισης σε 10 κράτη-μέλη έχουν εξεταστεί. Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία, Βέλγιο, Κροατία, Ιταλία, Λετωνία, Ουγγαρία και Πορτογαλία. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες σε κάποια κράτη-μέλη ε, ε, ε, κάποια κρατημέλη θεωρούν ότι κάποιες εκδίδουσες χώρες είναι ε, προβληματικές και δεν ανταποκρίνονται στα εντάλματα από τις χώρες αυτές και άλλοι περιμένουν να εξετάσουν κατά περίπτωση. Οπότε οι δικαστές πρέπει να σας πω ότι βασίζονται στα κρατη σε διάφορες πηγές. Κάποιοι λαμβάνονται, λαμβάνουν υπόψη τα όσα λέει η CPT του, του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συνθήκες και άλλοι βασίζονται σε άρθρα στις εφημερίδες ή σε ΜΚΟ που περιγράφουν συνθήκες ε, κράτησης. Προσπαθήσαμε την τελευταία χρονιά να περάσουμε ε, σε μια νέα εποχή και να ζητήσουμε από τον οργανισμό στη Βιέννη, από την Επιτροπή εκεί, να θεωρείται ως ο βασικός σταθμός επικοινωνίας που θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων και στην οποία θα μπορούν να στραφούν όλες οι δικαστικές αρχές. Δημιουργήθηκε το 2019 και σε ένα τόπο μπορούμε να βρούμε ε, πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν βαθμολογεί ε, αλλά περιγράφει ε, το πώς είναι οι συνδίκες κράτησης, το κατά πόσο έχουν πρόσβαση ε, σε, σε περίθαλψη, τις υγειονομικές συνθήκες και το κατά πόσο είναι ευάλωτοι σε βία περιστατικά οι κρατούμενοι. Οπότε αυτό είναι καλό. Για τις συνθήκες κράτησης μου υπενθυμίζει ότι υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα με την εφαρμογή που είναι η διάρκεια της πρώτης δίκης κράτησης. Αυτό αναφέρθηκε και ε, στην, ε, ε, στο δικό σας ψήφισμα. Γιατί συνήθως το 20% του πληθυσμού στα σοφρονιστικά καταστήματα είναι σε αναμονή δίκης. Σε κάποια κράτη είναι μόνο μερικοί μήνες αυτή η διαδικασία και σε κάποιους μένουν χρόνια φυλακή πριν δικαστούν η DG Justice έκανε μία ε, ε, συγκριτική μελέτη, την οποία τελειώσαμε το 2006, και τα κράτη-μέλη σε μεγάλο βαθμό ε, συμφωνούν ε, με και συμμορφώνονται με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και με τις αποφάσεις του, του Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Η κυρία Γιουρόβα δεν έχει προτείνει ακόμα νομοθεσία, γιατί, γιατί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και εξαιρετικά σύνθετο το θέμα αυτό της προδικαστικής κράτησης. Χρειάζεται καινοτόμες λύσεις εξυγχρονισμό, για παράδειγμα, των ε, ε, ποινικών ε, κωδίκων στα κράτη-μέλη, όπως επίσης και σε ενίσχυση του δικαστικού σώματος. Δεν αποκλείεται η νέα επίτροπος, ο κύριος Ρέινιετς συγκεκριμένα, να εξετάσει πιο λεπτομερώς τα θέματα αυτά και να προτείνει κάποια μέτρα. Τώρα μπορώ να περάσω στο τελευταίο προβληματικό θέμα που είναι το διπλό αξιόπινο είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει ε, πολλές φορές για τον κύριο Πουτσμόν. Και εδώ έχουμε ένα κατάλογο δικημάτων για τον οποίο δεν έχει ελεγχθεί ε, ε, το διπλό αξιόπινο, θα πρέπει να διευρυνθεί. Όταν λοιπόν συζητάμε το θέμα αυτό με τους νομικούς, με δικαστές και με εισαγγελείς, τα προβλήματα δεν μοιάζουν να είναι τόσο πολύ για το ότι κάποια δικήματα όπως η στάση για παράδειγμα δεν συμπεριλαμβάνονται ε, στον κατάλογο για τον οποίο δεν ισχύει ο έλεγχος του διπλού αξιόπινου. Ο κατάλογος αυτός μπορεί σύμφωνα με την απόφαση της Κούρια να διευρυνθεί και με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου. Αλλά δεν είχαμε ποτέ ε, κάποιο τέτοιο αίτημα. Έχουμε στο άρθρο 2.2 ένα κατάλογο αδικημάτων που περιγράφονται με αρκετά αόριστο τρόπο, δηλαδή απάτη, σαμποτάζ, το οποίο έχει δεχθεί πάρα πολλές ερμηνείες και πολύ συχνά τα εντάλματα εκδίδονται για αδικημένα τα οποία δεν είναι καν ποινικό αδίκημα στο άλλο κράτος μέλος. Δηλαδή απάτη με μικρή ζημία μπορεί να είναι ε, ποινικό αδίκημα ή όχι, στην οποία περίπτωση δεν εξετάζεται το διπλό αξιόπινο. Και τέλος, και ίσως αυτό σας ενδιαφέρει, είναι ο σχεδιασμός της αναθεώρησης του εντάλματος αυτό και της σχετικής απόφασης πλαίσιο. Η προηγούμενη Επιτροπή είχε ε, δηλώσει πως δεν είχε σκοπό να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση και μέχρι στιγμής η πλειοψηφία των κρατών μελών ήταν κατά του να ξανανοίξουν την απόφαση πλαίσιο. Γιατί ε, κυρίως φοβούνται πως θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και η αποτελεσματικότητα του εργαλείου ενδεχομένως θα πολεστεί. Θα ήταν δύσκολο λοιπόν να βρούμε ένα νομικό συμβιβασμό για να εξισορροπήσουμε μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αμοιβέ εμπιστοσύνη. Και το έχουμε δει αυτό με τη δίμευση ε, των περιουσιακών στοιχείων, ε, τι έγινε με το σχετικό κανονισμό. Οπότε δεν θα έπρεπε να αφήνουμε το ΔΕΚ ε, να αναλαμβάνει το ρόλο του νομοθέτη, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά με την ομολογία που τρέχει συνέχεια. Οπότε, το να ξανανοίξουμε όπως ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημαίνει νέα οδηγία, ε, νέες συζητήσεις για όλες τις διατάξεις και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πως θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί πριν ε, ανοίξουμε αυτό το ενδεχόμενο για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που σας πίεσα λίγο, αλλά ε, χρειαζόταν αυτή η πίεση διότι θα πρέπει να υπάρχει χρόνος και η συζήτηση. Ο, το λόγο έχει ο κύριος Χιμένες Βιγιαρέχο, μέλος της ομάδας της Eurojust για τα μέσα δικαστικής συνεργασίας και εθνικό μέλος για την Ισπανία. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι προηγούμενες παρεμβάσεις ήταν τόσο λεπτομεριακές που καθιστούν το έργο μου πολύ πιο εύκολο. Θα μιλήσω δηλαδή όχι μόνο για νομικά αλλά και για πρακτικά θέματα. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα μέσον που χρησιμοποιείται ευρέως 150.000 εντάλματα σύλληψης ε, έχουν εκδοθεί μεταξύ το, 2005 και 2006 και πάνω από 43.000 εντάλματα σύλληψης έχουν εκτελεστεί. Είναι λοιπόν το πιο επιτυχές μέσον μπορώ να πω μέχρι τώρα. Όμως υφίστανται θέματα γιατί υπάρχουν πολλές προκλήσεις ως προς την χρήση αυτού του δικαστικού μέσου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, ε, δόθηκε μια μεγάλη μάχη για την χρήση αυτού του μέσου τα τελευταία χρόνια. Η Eurojust ε, προβάλλει αυτή την δικαστική διαδικασία, ιδιαίτερα για θέματα ποινικού δικαίου. Έχουμε εκδώσει πολλές εκθέσεις ως προς το θέμα της αναλογικότητας για το πώς μπορούμε να επιλέξουμε το δικαστικό μέσο, το ε, πιο προσήκον δικαστικό μέσο. Είχαμε ε, μία ε, έκθεση, εκδώσαμε μία έκθεση το 2014 μετά εκδώσαμε ε, και μία έκθεση ως προς το, τα πρακτικά ζητήματα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και τις ε, περιπτώσεις παράδοσης μεταξύ 14-16 και τώρα αναθεωρούμε ε, αυτό το πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο από το 17 μέχρι το 19 και μέχρι το τέλος του έτους θα δημοσιευτεί αυτή η έκθεση. Η συζήτηση αυτή είναι άκρος επίκαιρη και για εμάς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και πολλές εξελίξεις. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι τα θετικά και τα αρνητικά και τα σκιώδη δηλαδή σημεία του εντάλματος σύλληψης και ε, οι ελλείψεις και τα χάσματα δεν οφείλονται στην απόφαση πλαίσιο, αλλά επειδή δεν υπάρχει ε, ισόρροπη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακολουθεί το ζήτημα για πολύ καιρό και είναι σε καλύτερη θέση να προβεί σε μια αξιολόγηση σε σχέση με εμένα, ότι παρουσιάζει μια έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί πριν από το καλοκαίρι φέτος σε σχέση με την ε, εφαρμογή αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Η Επιτροπή βρίσκεται στην καλύτερη θέση να το κάνει αυτό, αλλά από πρακτικής πλευράς ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συμβουλευτικές διαδικασίες που εντάσσονται στην απόφαση πλαίσιο, αλλά και στα δικαστικά μέσα αναγνώρισης, αμοιβέ αναγνώρισης. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να εκινήσει μία διαδικασία ε, ε, διαβούλευσης. Υπάρχει και ο χρυσός κανόνας της αμοιβαίας αναγνώρισης της δικαστικής συνεργασίας, αλλά δεν ε, λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή δεν ε, αντλεί κανείς από αυτά τα προτερήματα για, για να τα χρησιμοποιήσει πάντα, ιδιαίτερα ως προς την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Εάν λάβουμε υπόψη την δικαστική φύση αυτού του μέσου. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι το ένταλμα σύλληψη σε σχέση με άλλα θέματα αμοιβές αναγνώρισης ε, είναι, έχει ένα διμερές πλαίσιο και όχι πολυμερές. Όπως ε, και το γεγονός ότι οι εθνικές δικαστικές ε, αρχές ακολουθούν μία επιταχυμένη επιταχυνόμενη διαδικασία και γι' αυτό αυτό θα μειώσει, τις, ίσως θα μείωνε τις εργασίες της Eurojust, αλλά αυτό δεν ισχύει, γιατί οι ανοιχτές περιπτώσεις αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Και αν συγκρίνουμε τα στοιχεία με το 18 είχαμε 442 υποθέσεις, ε, διμερείς υποθέσεις που σχετίζονται με με τη βελτίωση της κατάστασης ως προς τα ε, εντάλματα σύλληψης. Πέρσι όμως είχαμε 599 υποθέσεις και τα αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν την ανάγκη ε, αρρωγής και εξειδικευμένων συμβουλών ως προς αυτές τις υποθέσεις. Ε, η Eurojust χρησιμοποιεί την ε, απόφαση πλαίσιο ως μέσον επίλυσης διαφορών και δυνάμει του άρθρου 16.2 της απόφασης αυτής πλαισίου χρησιμοποιούμε αυτό το πλαίσιο για την δική μας ε, νομολογία και η κατευθυντήριες γραμμές έχουν αναθεωρηθεί, αναθεωρήθηκαν το 2019 και υπάρχει και μία διάταξη στο άρθρο 17 σε σχέση με τις παραβιάσεις, τη μη τήρηση προθεσμιών αλλά ο νέος κανονισμός μας δίνει τη δυνατότητα να συνδράμουμε ως διευκολυντές, διότι στο άρθρο 2.2 αυτού του νέου κανονισμού ε, δυνάμει του πρώην άρθρου 3 της απόφασης της ε, Eurojust, η Eurojust διευκολύνει την δικαστική συνεργασία ιδιαίτερα ως προς την αμοιβαία αναγνώριση και τις σχετικές αποφάσεις. Υπάρχει λοιπόν νομική βάση για την ε, παρέμβασή μας, αλλά κάθε φορά που υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης, η Eurojust θα μπορούσε να συνδράμει τις εθνικές αρχές γιατί είμαστε ένα δικαστικό φόρουμ για διάλογο. Μπορώ να σας μιλήσω και για απτά παραδείγματα πιο, συχνά, οι πιο συχνές υποθέσεις, η πρώτη ομάδα υποθέσεων αφορά αίτημα επιπρόσθετης πληροφόρησης. Έχουμε πολλά, πολλές τέτοιες αιτήσει δυνάμει του άρθρου 15 της απόφασης και αυτή είναι μία από τις ε, σημαντικές μας ε, προκλήσεις Επίσης, μιλάμε για επιπρόσθετες πληροφορίες όταν οι εθνικές ε, δικαστικές αρχές τις χρειάζονται και όταν έχει, δεν έχει ε, ληφθεί απόφαση σε μια προγενέστερη υπόθεση. Οπότε εμείς θα να υποστηρίξουμε τις εθνικές ε, δικαστικές αρχές. Επίσης, ε, ζητούνται διασαφηνίσεις από τις εθνικές ε, δικαστικές αρχές μέσα σε μέρες ή ώρες, διότι η ίδια, το ίδιο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι μια κατεπίγουσα διαδικασία όπως ορίζει το άρθρο 17.1 της απόφασης πλαισίου τα αιτήματα αυτά αφορούν την ταυτοποίηση του, του φυσικού προσώπου και έχουμε υπόψη συγκεκριμένες ε, υποθέσεις, γνωστές υποθέσεις και φυσικά και το ε, εθνικά ζητούνται και τα εθνικά εντάλματα σύλληψης, η περιγραφή του αξιόπινου, ε, και θέματα ε, του διπλού αξιόπινου με βάση και την εθνική, το εθνικό ένταλμα σύλληψης για να δούμε την φύση αυτών των, ε, της διακαστικής συνεργασίας και φυσικά και πληροφορίες τύπου follow-up μετά τη, ε, τις διαδικασίες παράδοσης σε συγκεκριμένες εγγυήσεις σε σχέση με την ερήμην καταδίκη προσώπων και ε, το άρθρο 27.4 σχετίζεται με την ε, αρχή της εξειδίκευσης η οποία προαπαιτείται εδώ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η νομολογία του ιδιαίτερα σε σχέση με το τη δίκαιη δίκη, τις συνθήκες φυλάκισης, την ερημοδικία και ούτω καθεξής. Ε, εδώ και σε τέτοιες περιπτώσεις ζητούνται επιπρόσθετες πληροφορίες και αυτό που έχει σημασία είναι τι είναι αναγκαίο και τι είναι προσήκον, τι είναι σχετικό με την υπόθεση. Και η πραγματική πρόκληση με βάση την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι να βρει η Eurojust τη σωστή ισορροπία μεταξύ των των πληροφοριών και των προθεσμιών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σωστό feedback σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές για να συμμορφωθούμε με την πρόσφατη ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η ε, δεύτερη ομάδα ε, πρακτικών ζητημάτων που, που ανακύπτουν αφορούν τις, ε, τα θέματα μη αναγνώρισης. Δηλαδή πότε ισχύει η μη αναγνώριση για την εφαρμογή αποφάσεων των δικαστικών αρχών και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο τηρούνται τα προαπαιτούμενα ή όχι. Και αυτό που έχει σημασία είναι σε σχέση με διώξεις κατά πόσο και η ε, Eurojust συλλέγει όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις ε, υποθέσεις για να ληφθούν αποφάσεις ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως το non bis in και να μπορέσουμε να συνδράμουμε τις εθνικές δικαστικές αρχές για να μπορέσουν να αποφανθούν και αυτό που έχει σημασία είναι ποιο είναι το κράτος εκτέλεσης της απόφασης. Πολλές φορές έχουμε ε, υποθέσεις διπλού αξιόπινου, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θέματα διπλού αξιόπινου σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζονται με το, με το αξιόπινο των πράξεων και με συγκεκριμένα αδικήματα που δεν σχετίζονται πάντα με την εργασία της Eurojust. Έχουμε και ε, θέματα για το πόσο μπορούμε να συντονίσουμε τις εργασίες του εντάλματος με την Ευρωπαϊκή ε, Διαταγή Επίβλεψης και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας δυνάμει των άρθρων 22 και 25 σε περιπτώσεις που έχουν αναβληθεί οι παραδόσεις για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους. Και βεβαίως οι επιπτώσεις της νομολογίας. Εκεί αποτιμούμε τις αποφάσεις, ε, ε, αποφάσεις Αρανιώση και Καλδαράρου και έχουμε και μία θεματική πτυχή. Γιατί το 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σε σημαντικές υποθέσεις, όπως τις 27 Μαΐου 2019 που είχε μεγάλες επιπτώσεις ως προς την συνεργασία των δικαστικών αρχών και η Eurojust έκδωσε ένα ερωτηματολόγιο για μια χαρτογράφηση των γενικών εισαγγελιών για να δούμε κατά πόσο οι εισαγγελικές αρχές μπορούν να εκδώσουν ένα ένταλμα, σύλληψης και ε, για να κρίνουμε την ε, ανεξαρτησία του δικαστικού. Ε, ως προς ε, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, μία άλλη σειρά αποφάσεων, προθήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για πραγματική δικαστική προστασία και τώρα ενημερώνουμε αυτά τα στοιχεία. Για να συμπεράνω θα ήθελα ένα λεπτό για να ε, τονίσω ότι σε έναν ιδεατό κόσμο αμοιβαία αναγνώρισης ε, ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία αναγνώριση ή ε, μη αντιμετώπιση άλλων συναφών ζητημάτων. Σε έναν ιδεατό κόσμο δηλαδή, οι δικαστικές αρχές επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους. Αλλά εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε ως Eurojust τις δικαστικές αρχές, ιδιαίτερα όταν ζητούν επιπρόσθετες πληροφορίες και με βάση την πρόσφατη νομολογία του, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Eurojust ε, συνδράμει σημαντικά για τη χρήση αυτού του μέσου και φτάσαμε σε πολλές περιπτώσεις σε μία λύση συμμόρφωσης, γιατί ακολουθούμε την δικαστική διαδικασία και πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε αυτό το τομέα έχουμε συνδράμει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ, όλους τους ομιλητές. Πραγματικά τιμάτε την Επιτροπή μας που ήρθατε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας, την εμπειρία σας και ζητούμε συγγνώμη για την πίεση. Και πάντα έχουμε χρονική πίεση εδώ. Αλλά θα πρέπει να αρχίσει η συζήτηση. Ακούμε πρώτα τους σκιώδες. Πρέπει να ακούσουμε τις απόψεις των σκιωδών Πρώτος ο κύριος Φράνκο Ρομπέρτη, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Δύο λεπτά αν μπορείτε, θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Σε δύο λεπτά δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Σήμερα έχουμε την απτή απόδειξη της σημασίας αυτού του δικαστικού μέσου. Εγώ υπήρξα μάρτυρας της χρήσης αυτού του μέσου και αυτό το βλέπουμε και με την άξιση της ε, νομολογίας και στην εσωτερική ενόμη τάξη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και γι' αυτό χτες είπα στον Επίτροπο Σχοινά ότι λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί έγιναν σοβαρές περικοπές στη χρηματοδότηση της Eurojust. Εγώ προβλέπω ότι στα επόμενα χρόνια θα ε, έχουμε μία φθήνουσα ε, χρηματοδότηση και συνεργασία μεταξύ δικαστικών αρχών γιατί μειώνεται και ο ρόλος της Eurojust. Σας ευχαριστώ για αυτές τις εισηγήσει, γιατί πέρα από τα στατιστικά στοιχεία που μας έδωσε και η εκπρόσωπος της Επιτροπής, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ζητήματα αρχής, γιατί μιλάμε για την εναρμόνιση των δικαστικών μέσων. Άρα θα πρέπει να ορίσουμε τη συνεργασία των δικαστικών αρχών και η Ευρωπαϊκή ε, οι Ευρωπαϊκές Αρχές και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Θα πρέπει λοιπόν να ε, βλέπουμε αν υπάρχει πραγματική ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση της Πολωνίας. Άρα η όλη αρχή αδειοδότησης θα πρέπει να εγκρίνεται από μία ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή από ένα δικαστήριο. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε το, τα θέματα συμμόρφωσης ως προς το κράτος εκτέλεσης και βεβαίως και τις συνθήκες κράτησης. Επίσης, το άρθρο 2 αναφέρεται σε 22 είδη αδικημάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να προσπαθήσουμε να ορίσουμε τα αδικήματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα και τα σχετικά. Θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς διότι αυτό είναι ύψη της σημασίας για να ορίσουμε αυτά τα εγκλήματα. Υπάρχουν και άλλα αδικήματα που έχουν ανακύψει τα τελευταία 18 χρόνια, ε, δηλαδή τη μαύρη εργασία, την δουλεμπορία, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και ούτω καθεξής. Είμαι πολύ αισιόδοξο ως προς τη δυνατότητα βελτίωσης ε, της εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης που να υπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστούμε κύριε Ρομπέρτη. Είπατε πολλά, καλύψατε πολλά σε δύο λεπτά και κάτι. αλλά είπατε θέματα, αναφερθήκατε σε θέματα ουσίας και σας ευχαριστούμε αυτό. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε μεγάλη πίεση χρόνου. Θα περάσουμε στον επόμενο σκιώδη, που είναι η κυρία Μαϊτέ Ορτοντουά. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και εγώ να έχει περισσότερους πόρους οικονομικούς η Eurojust, γιατί έχει τεράστιο φόρτο εργασίας, γιατί ζούμε στο χώρο Σέγγεν. Ε, και στην παγκοσμιοποίηση είναι πολύ μεγαλύτερες ε, οι δυνατότητες ε, τέλες αξιόπιων πράξεων και το διεθνές έγκλημα. Πήγαμε στη Eurojust και μας παρουσίασαν μια υπόθεση που είχαμε δολοφονίες, ξέπλυμα χρήματος, λαθρεμπόριο ναρκωτικών στα κράτη-μέλη με ανθρώπους που είχαν πολλές ηθαγένειες. Ε, ότι κάποιος σκότωσε από το κράτος Α, σκότωσε κάποιος στο κράτος Β και τα λοιπά και είχαμε διάφορες ηθαγένειες και υπηκότητες. Και επίσης σχεδίαζαν και κοιτούσαν και τι ώρα άνοιγαν οι τράπεζες για να ε, ε, νομιμοποιήσουν τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες και θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο περίπλοκη κατάσταση εάν ε, κάποιο είχε διπλή ηθαγένεια με κάποιο κράτος μη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει κίνδυνο ατιμορρησία. Πραγματικά σε αυτή την κατάσταση ζούμε στη χώρα Σέγγεν που έχουμε ελευθερία κινήσεων και κυκλοφορία, αλλά υπάρχουν τεράστιε ακόμα δυνατότητες για τα σημεία που ακόμα δεν έχουν καλυφθεί ή ε, χωλένουν στην ε, αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Είμαστε στο Σέγγεν πλέον και ε, είναι νέε οι ανάγκε, έχει αλλάξει ο κόσμος. Ακούσαμε για αυτές τις συγκεχημένες και θολές κατηγορίες που φυσικά θα πρέπει να επαναορίσουμε και να διευκρινίσουμε και αν δεν υπάρξει καλύτερη ε, συνεργασία και συντονισμός πρέπει να ορίσουμε καλύτερα και το λέω στη δεύτερη ε, ομιλήτρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα αυτά τα θέματα δεν είναι πολιτικά ουσιαστικά, τεχνικά είναι. Και τα δεδομένα, γιατί βλέπουμε το 2017 έχουν εκδοθεί 17.491 εντάλματα και γύρω στις 6.000 εκτελούνται, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τι έγινε, γιατί δεν είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να διαβιβάζουν ε, και δεν ξέρουμε πόσοι είναι φυγάδες, φυγόδικοι και πόσοι δεν έχουν ε, εντοπιστεί. Πάνω από 10.000 εντάλματα δεν εκτελούνται. Καταλαβαίνεις την απογοήτευση, τη ματέωση και των δικαστικών και των Ευρωπαίων πολιτών που θα σταματήσουν να εμπιστεύονται το σύστημα το θέμα της εμπιστοσύνης στο σύστημα δεν είναι θέμα πολιτικής εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών που τόσο πολύ φοβάται το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι και ένα θέμα εμπιστοσύνης των πολιτών στο δημοκρατικό σύστημα και στο δικαστικό σύστημα. Και αν εμείς τρομάζουμε και δηλιάζουμε και δεν θέλουμε να κάνουμε καμία αλλαγή, αθετούμε ε, μία από τις ε, βασικέ υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του να εμπιστεύονται οι πολίτες τι δημοκρατίε τους. Λέω λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο να εμπιστεύεστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δίνετε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Όλα αυτά που ακούσαμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτέ οι βελτιώσει οι περισσότερε. δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά, Αμυγό τεχνικά. Δεν ανοίγουμε κανένα σκότου αιώλου. Τη δουλειά μα θέλουμε να κάνουμε υπεύθυνα άλλο θέμα. Φόβους. Ε, μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη και αγωνίες για άλλα θέματα. Αλλά γι' αυτό που εμείς μπορούμε να ε, επιτύχουμε με αυτό το ε, μέσο της δικαστικής συνεργασίας, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τίποτα, ούτε να κρυβόμαστε. Όλα αυτά τα στοιχεία που ακούσαμε μας δείχνουν ότι μπορεί να βελτιωθεί αυτό το μέσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παγάσα Ορτούντουα. Από τους Πρασίνους. Η κυρία Ντελμπό Σκορφίλ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε. Ε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Αλλά τον Ιούνιο θα φέρει ε, τις προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο επίσης εργάζεται. Ε, για ε, το άρθρο 17 γίνεται μια αξιολόγηση σε όλα τα κράτη-μέλη, έχει αρχίσει και θα τελειώσει το 2021. Ήθελα να το πω αυτό εισαγωγικά για να εξηγήσω ότι βεβαίως θα πρέπει να κοιτάξουμε την εφαρμογή, αλλά όχι βεβαιασμένα για να αλλάξουμε οπωσδήποτε κάτι. Πρέπει να δούμε όλες τις αξιολογήσεις που γίνονται από διάφορα θεσμικά όργανα πριν αρχίσουμε ή πριν συνεχίσουμε τις αλλαγές. Αυτό είναι το πρώτο. Um, Οι περισσότεροι το είπατε, αλλά ε, θα πρέπει ε, να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στη δίωξη και τα δικαιώματα της υπεράσπισης. Δεν να σας άκουσα, αλλά δεν ξέρω, μπορεί ε, να παράξω γιατί δεν τα ακούμε και όλα. Δεν σας άκουσα να λέτε πολλά πράγματα για την εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και των δικηγόρων εξ όσων κατάλαβα, γιατί είμαι και πάρα πολύ καινούργια σε αυτά τα θέματα, είναι ζήτημα και μείζον. Θα πρέπει όλοι στην Ευρώπη να έχουν αντίστοιχη εκπαίδευση και να έχουν και εκπαίδευση στο να κατανοούν ο ένας τον άλλον και όλα αυτά τα διαδικαστικά θέματα και τα δικονομικά. Θέλω να ακούσω περισσότερες λεπτομέρειες για την ουσιαστική υπεράσπιση Γιατί καμιά φορά οι συνηγοροί δεν έχουν πλήρη ε, πρόσβαση ε, στη δικογραφία. Υπάρχει το θέμα της χώρας που εκδίδει και της χώρας που εκτελεί, ε, θέμα δικαιωμάτων, θέματα μεταφράσεων, κατανοούν πάντα τα δικαιώματά τους. Και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις. Γιατί προς το παρόν δεν πιστεύω ότι ε, ε, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα δώσει χρήματα τώρα στα κράτη-μέλη για τις φυλακές. Πώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης. Τι γίνεται με το δικαίωμα στην έφεση και στη χώρα που εκδίδει και στη χώρα που εκτελεί το ένταλμα. Μιλήσατε για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ενέχεται και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Θα ήθελα λίγο περισσότερες πληροφορίες το είπε και η προλαλήσασα, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των ενταλμάτων που εκδίδονται και εκείνων που εκτελούνται. Έχω την τάση να πιστεύω ότι αυτό γίνεται ε, γιατί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους τα κράτη-μέλη. Αλλά μπορεί να γίνονται και πολλά λάθη στην έκδοση αυτών των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Εσείς αυτό πώς το αξιολογείτε. Γίνεται κακή χρήση του εργαλείου αυτού Μήπω δεν εκδίδονται πάντα με σωστό τρόπο τα εντάλματα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει το μικρόφωνο ο Πρόεδρος. Ο κύριο Μπουξαντέ από το ΙΣΙΑ. Gracias, gracias presidente y Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όσους έχουν πάρει το λόγο και σίγουρα θα μπορέσουμε να ζητήσουμε περισσότερες μελέτες, αλλά το βασικό είναι έχοντας ακούσει τους τρεις ε, εισηγητές και έχοντας αναγνώσει το έγγραφο εργασίας της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 28 Αυγούστου 2019, είναι κάποια θέματα τα οποία ε, τα έχουμε κατανοήσει, τα έχουμε συμφωνήσει και θα πρέπει για αυτά να πούμε κάτι παραπάνω το ένταλμα είναι πετυχημένο. Έχει αυξηθεί ε, ο αριθμό αιτήσεων και αυτό αποδεικνύει πω οι δικαστικέ αρχέ των κρατών μελών ενδιαφέρονται μέσω αυτού να ζητούν τη συνεργασία άλλων δικαστικών δικαιοδικουσιών. Όμως δεν είναι πραγματική αυτή η επιτυχία, γιατί όταν είναι 70% ε, τα αιτήματα αυτά τα οποία παραμένουν εκτελεστά τότε δημιουργούνται ερωτηματικά. Επίσης, φαίνεται πως οι ίδιοι οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τις ελλείψεις του ευρωπαϊκού εντάλματος για να αποφύγουν ε, το χέρι της δικαιοσύνης, προσφεύγοντας λοιπόν σε διασυνοριακή δράση, κάτι το οποίο απαιτεί από εμά μία απόκριση, γιατί πολύ συχνά χάνουμε ε, τον καιρό μας με γενικές δηλώσεις εμείς ως πολιτικοί και ξεχνάμε πως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και το δικαίωμα του θύματος γιατί το σύγχρονο δίκαιο θα πρέπει να έχει ως στόχο την ικανοποίηση του θύματος. Εδώ και 200 χρόνια μιλάμε μόνο ε, για την προστασία του ενδεχόμενου υπόπτου. Πρώτα απ' όλα, υποχρέωση να στέλνονται πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, η ανάγκη να στήσουμε εργαλεία τα οποία ε, στο κράτος υποδοχής ε, τέτοιου είδους αιτήματο να ανταποκριθεί ε, και εφόσον αποδειχθεί ότι απέρριψε το αίτημα αυτό χωρίς αιτία να υπάρχει κάποιος μηχανισμός επιβολής συμμόρφωσης. Και για τον ορισμό των αδικημάτων και τα 32 που βρίσκονται στον κατάλογο. Ίσως θα έπρεπε να δούμε και πιο συγκεκριμένους ορισμούς ή ε, να πούμε ε, στο αξιόπινο το οποίο σημαίνει πως θα ακολουθήσουμε ε, το δικαίωμα στην προστασία που ακολουθούν όλα τα κράτη-μέλη και να ενισχύσουμε ε, ότι βοηθά ε, τον δικαστή να αποφασίσει χωρίς να χρησιμοποιήσει τη δικριτική του ευχέρεια. Αυτό το κομμάτι θα πρέπει να περιορίσουμε γιατί τα προβλήματα ε, προκύπτουν. Πρώτον, όταν ο, στο κράτος υποδοχής ο δικαστής αξιολογεί το διπλό αξιόπινο, αυτό πρέπει να το εκφράσουμε συγκεκριμένα έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα διακριτικής εφαρμογής και να είναι πολύ σαφής ο κατάλογος και ευρύς ε, των ε, αδικημάτων που ε, εμπίπτουν στο διπλό αξιόπινο και δεύτερον να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στο πώς αξιολογούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όχι να αφήνουμε τους δικαστές να διαβάζουν άρθρα σε εφημερίδες για να το αποφασίσουν, να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος. Και ξέρουμε και την υπόθεση Χαουρέδιου που δικάστηκε το βελγικό κράτος ε, γιατί έκρινε ε, πως στην ε, Ισπανία δεν γίνονται σεβαστά τα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αντίστροφα ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να απαντήσει πως στο Βέλγιο δεν συμβαίνει αυτό. Η κυρία Ντέλη από την ΚΟΕ γιατί είναι και η, η Με συγχωρείτε που βγήκα ε, στη μέση της παρέμβασης. Δεν ήταν έλλειψη σεβασμού προς Απλώς δεν μπορώ ακόμα να είμαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Λοιπόν, από τις πληροφορίες που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017, 109 εντάλματα απορρίφθηκαν βασιζόμενοι σε, με αιτιολόγηση τα ε, θεμελιώδη, ε, δικαιώματα. έχουμε στοιχεία για το ποια θεμελιώδη ε, δικαιώματα επικαλέστηκαν. Έχουμε τέτοιου είδους στοιχεία πόσες περιπτώσεις απορρίφθηκαν λόγω διπλού αξιόπινου. Και από αυτά τα στοιχεία ίσως να προκύψουν και κάποιες πληροφορίες για το είδος των υποθέσεων που απορρίφθηκαν ε, γι' αυτό το λόγο. Γιατί ίσως υπάρχουν βασικοί λόγοι για την απόρριψη με θελημιώδη δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε εμείς να παρακολουθούμε. Και αυτό ίσως ε, να ενημερώσει και τις συζητήσεις μας όταν μπούμε ε, σε εκείνο το θέμα. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι προηγούμενοι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το θέμα αυτό μεμονωμένα. Θα πρέπει να δούμε και τις ε, συναρτώμενες οδηγίες η πρόσβαση σε ε, δική δικηγόρο, ε, η το επίδομα παινίας, το επιδότημα παινίας ε, και όλα τα σχετικά για τα θέματα τα οποία ε, προκύπτουν και τα οποία προστατεύονται ατελώς σε πολλές υποθέσεις. Για να δούμε λοιπόν, εφαρμόζονται σωστά όλες οι σχετικές οδηγίες, γιατί οποιαδήποτε τέτοια ε, προβληματική εφαρμογή μπορεί να παραβιάζει και άλλα δικαιώματα που βρίσκονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και όχι μόνο αυτό του αξιόπινου ή του δεδικασμένου. Επίσης, τι γίνεται όταν έχει εκδοθεί ένταλμα σε προς δύο ε, διαφορετικές χώρες. Στην περίπτωση αυτή τι υπερισχύει και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βασιστεί στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στην ομολογία σχετικά με το οι διώκουσες αρχές να μην εκτελέσουν το ευρωπαϊκό ένταλμα λόγω παραβιάσεως των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και μέχρι να θεωρήσουμε το ένταλμα, μέχρι να λάβουμε υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα, μήπως θα έπρεπε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, ή να περιορίσουμε τη χρήση του έτσι ώστε ε, να το αποφασίσουμε όταν και τα υπόλοιπα κομμάτια έχουν βρει τη θέση τους. Α, οκ, okay, τελειώσαμε με τους σκιωδές, αλλά έχουμε και κάποια μέλη τα οποία θέλουν να λάβουν το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι και θα ξεκινήσουμε. Ο κύριος Κινίτσι και μετά εσείς. Τα παρόλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκαλεσμένους μας για τις εισηγήσει που είναι άκρος ενδιαφέρουσε στο θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Είναι το πιο σημαντικό μέσο δικαστικής συνεργασίας. Επειδή και εγώ προέρχομαι από το δικαστικό τομέα, δίνω ε, μεγάλη σημασία στη δικαστική αυτή συνεργασία. Γι' αυτό θα σταθώ στο άρθρο 2 που προβλέπει ε, θέματα αξιόπινου όταν μιλάμε ιδιαίτερα για το διπλό αξιόπινο. Τα θέματα αυτά επικαιροποιούνται και αλλάζουν και οι μορφές εγκληματικότητας. Και εδώ μιλώ για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για το, την απόφαση πλαίσιο και που δεν έχει οδηγήσει στην εναρμόνιση των νομοθεσιών. Νομίζω ότι η εναρμόνιση των νομοθεσιών έχει μεγάλη σημασία για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μέλων. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο δεν κρίνεται ότι ήρθε η στιγμή για να αλλάξουν αυτοί οι ορισμοί για να προσαρμοστούν στην ε, πραγματικότητα ως προς εγκληματικές δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το άρθρο 647α και το άρθρο 416 αντίστοιχα του Ισπανικού και του Ιταλικού ποινικού δικαίου αναφέρονται σε βελτίωση του εντάλματος σύλληψης η εκπρόσωπη της Επιτροπής μίλησε για τις συνθήκες κράτησης και το θέμα αυτό ανέκυψε ακριβώς επειδή οι φυλακές ε, ξεχυλίζουν από κρατούμενους. Ε, και όπως είπε και ο συνάδελφος Ρομπέρτη, αναρωτιέμαι κατά πόσο δεν θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μια γενικότερη βελτίωση και να υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές για τις ε, συνθήκες κράτησης. Και εγώ θεωρώ ότι η Eurojust ε, στην ουσία μπορεί να διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να έχει την ε, κατάλληλη χρηματοδότηση. Δεν πρέπει να μειώνεται δηλαδή η χρηματοδότηση της Eurojust. Με συγχωρείτε που θα πρέπει να αποχωρήσω σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέει η κυρία Κέμπα. Θέλω να ευχαριστήσω ε, πολύ τους ομιλητές. Ήταν καταπληκτικές και οι ομιλίες σας και η συζήτηση. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ε, όταν ε, μεταφέραμε στην εθνική μας νομοθεσία το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη στην Πολωνία. Ήταν πολύ εντονή συζήτηση και είχαμε τη φιλοδοξία να είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και δεν σφάλαμε. Ε, είναι γεγονό. Μπορεί να έχει κάποιες ελλείψεις και προβλήματα αυτό το νομικό εργαλείο, αλλά θα άξιζε τον κόπο να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο γιατί αποδίδει. Ε, δανειζόμενοι από τις εμπειρίες, να βελτιώσουμε περισσότερο ε, το εργαλείο αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες ε, των δικαστηρίων. Καλό είναι να μην αμφισβητούμε ο ένας τις αρμοδιότητες των δικαστηρίων του άλλου. Η ε, εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική ε, και η εμπιστοσύνη στα κράτη μας. Θα πρέπει να αγωνιστούμε πολύ περισσότερο και πολύ πιο στεναρά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κατηγορίες αξιόπινων πράξεων και αναφέρομαι στους ομιλητές μας. Μήπως να το συζητήσουμε αυτό με τα κράτη-μέλη τι γίνεται με τα κομμουνιστικά εγκλήματα, για παράδειγμα. Δεν μπορεί ένα κράτος μέλος να αρνείται να εκδώσει ή να παραδώσει ε, κάποιον ε, στη χώρα όπου έχει εγκληματίσει. Έχουμε το παράδειγμα της ε, Σουηδίας, όπου έχει παραγραφεί ένα αδίκημα, το οποίο στην Πολωνία όμως δεν παραγράφεται. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιων ανθρώπων Και κάποιοι είχαν πάρει πολιτικές αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις με πολιτικά κριτήρια εις βάρος κάποιων άλλων και μελών των ενόπλων δυνάμεων και ε, τους προστατεύουν στη Σουηδία. Δεν τον εκδίδουν γιατί θεωρούν ότι έχει παραγραφεί. Ε, ε όμως ε, εγώ σας λέγω ότι στη συνεργασία των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη και να κοιτάει κανείς πότε παραγράφεται ε, ένα αδίκημα σε μια χώρα και πότε όχι. Εδώ έχουμε τρομακτικούς εγκληματίες, δεν μπορεί να γλιτώνουν τώρα για μένα ατιμόρυτοι. Ευχαριστώ. Ε, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ζητήσει κανένας άλλο το λόγο. Προτείνω, πριν δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας για να κλείσει, θέλετε να μιλήσετε κι εσείς, έτσι, να ακούσουμε όμως πρώτα τους ομιλητές στα μέλη του πάνελ για να απαντήσουν. The shadows and the rest of the members. Ακούσαμε τους ε, ομιλητές, κάνανε ερωτήσεις και οι σκιώδεις και οι υπόλοιποι. Μπορείτε ένα σύντομο σχόλιο για να απαντήσετε, να αντιδράσετε δίλεπτο έκαστος. Please. Thank you very much. So in two minutes I will try to take the questions all together. Θα να σας πω λοιπόν πως το πρώτο μας σχόλιο είναι μπορούμε να αξιολογήσουμε μόνο εφόσον υπάρχουν δεδομένα. Αν δεν στέλνουν τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε πλήρη εικόνα και δεν ξέρουμε πώς να τα αξιολογήσουμε. Δεύτερον, το ίδιο το εργαλείο Στη δεύτερη φάση της ε, αξιολόγησης θα κοιτάξουμε το κατά πόσο είναι συνεκτικό και βλέποντας το ευρωπαϊκό ένταλμα θα πρέπει να δούμε αν είναι ε, συνεκτικό με το διεθνές δίκαιο και επίσης με τον τρόπο που εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη, με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά και πώς ε, είναι διαδραστικό με το δικανικό και με το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών. Εξετάζοντας τα δεδομένα ε, του 2017 θα δείτε πως οι περισσότερα, πάρα πολλά εντάλματα ήταν για ε, ε, κλοπή και βλάβη ακίνητης περιουσίας. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο τούτο. Για τα δικανικά δικαιώματα και αν δούμε την Επιτροπή του 17 και για την πρόσβαση σε δικηγόρο, ε, τέσσερα κράτη-μέλη δεν έχουν καν ε, εφαρμόσει την οδηγία που λέει πως πρέπει να υπάρχει δικηγόρος στο, ε, πρόσβαση σε δικηγόρο στο κράτος έκδοσης. Και για τα θύματα στο εγχειρίδιο, εμεί έχουμε κάτι διαφορετικό από το ψήφισμα του 2014 και θα πρέπει ε, να εξετάζονται ε, τα ε, θύματα στην περίπτωση που θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν δικαιώματα του θύματος τα οποία θα πρέπει να προστατευτούν κατά τη διαδικασία. Διαδικαστικά δικαιώματα. Να ακούσουμε τώρα και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο λεπτά για να απαντήσετε. Καταρχήν, για τον κύριο Ρομπέρτη και τη σημασία της Eurojust συμφωνώ. Συμφωνώ, η αμοιβή εμπιστοσύνη ξεκινά με τις άμεσες επαφές μεταξύ των ε, επαγγελματιών του κλάδου. Θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Για το κατάλογο των 32 δικημάτων το είπα, συμφωνώ, υπερβολικά γενικό, γενικόλογος ο κατάλογος και για κάποια δήματα όπως το σαμποτάζ και την απάτη, καλό θα ήταν να έχουμε ένα πιο εναρμονισμένο ορισμό για να δούμε τι γίνεται με τα ε, εγκλήματα αυτά. Για τα στατιστικά, σας τα εξήγησα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των ε, εκδιδόμενων και των εκτελεσμένων ενταλμάτων, για αυτούς τους οποίους δεν μπορούμε να εντοπίσουμε, για παράδειγμα, τα πολλαπλά που έχουν ε, εκδοθεί για το ίδιο άτομο, εκτός από τις απόρριψεις, δηλαδή αν είναι άρθρο 4-6, τουλάχιστον εκτελείται η ποινή από το κράτος διαμονής. Για την εκπαίδευση των δικαστών, ναι, το εξετάζουμε. Έχουμε σεμινάρια συγκεκριμένα για τους δικαστές που είναι στο Ευρωπαϊκό ε, Δίκτυο, συγκεκριμένα σεμινάρια, αλλά έχουμε και άλλα σεμινάρια ανοιχτά σε ε, πολύ συναφείς κατηγορίες. Επίσης, μελέτες συμμόρφωσης, γίνονται γίνονται κράτη-μέλη και εξετάζουμε το κατά πόσο θα ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση για τις οδηγίες τούτες. Για την κατάχρηση αυτών των ενταλμάτων γνωρίζουμε πως μερικές φορές χρησιμοποιούνται με καταχρηστικό τρόπο, για παράδειγμα για την ανάκριση υπόπτων, αυτό με, την ευρωπαϊκή, ε, με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά αυτό έχει να κάνει για περιπτώσεις που μπορούν να εντοπιστούν μέσω του CIS εύκολα ε, τα άτομα αυτά ή αν μπορεί να τους παραδοθεί το ένταλμα ή η κλίση σε απολογία. Σε περίπτωση που έχουμε απόρριψη των ενταλμάτων λόγω ε, συνθήκων κράτησης, ίσως εκεί θα έπρεπε να έχουμε ένα νέο εργαλείο για παράδειγμα, να έχουμε μια μεταφορά της ε, διαδικασίας έτσι ώστε να μην επιτρέπουμε την ατιμορρησία. Θεμελιώδη δικαιώματα και τις ε, απορρίψεις στη Γερμανία, κυρία Ντέιλι, λόγω ε, κακών συνθήκων κράτησης στις εκδίδουσες χώρες και έχουμε περισσότερες καθυστερήσεις και απορρίψεις για το θέμα αυτό παρά για θέματα κράτους δικαίου η νομολογία όπως η περίπτωση Αρανιώζη και τα λοιπά προκύπτουν από ε, τέτοιου είδους αποφάσεις προσωρινές ε, Γερμανών δικαστών. Τι μπορούμε να κάνουμε. Όπως είπα και στην παρέμβασή μου έχουμε ήδη δημιουργήσει μαζί με την ε, υπηρεσία μια βάση δεδομένων έτσι ώστε οι επαγγελματίε του κλάδου να έχουν πρόσβαση στι πληροφορίες. Επίσης, στο θέμα της κράτη και των συνθήκων, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με ε, συνεργασία με ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης, δηλαδή χρηματοδούμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών ε, προληπτικών ε, υπηρεσιών, όπου σε εθνικό επίπεδο παρακολουθούνται από αυτού τους θεσμούς οι συνθήκες κράτησης, ε, συζητάνε διάφορες φορές και προσπαθούμε επίσης να βελτιώσουμε και την υποδομή των σοφρονιστικών καταστημάτων. Έχουμε κάνει ένα οδικό χάρτη του τι μπορούμε να κάνουμε με τα τρέχοντα ευρωπαϊκά κονδύλια και υπάρχουν δυνατότητες, Δηλαδή υπό τα διαστοτικά ταμεία, το ΕΤΠΑ, και επίσης με την ενεργειακή αποδοτικότητα. Κάποιες ε, φυλακές ε, στην Ουγγαρία ειδικά χρησιμοποίησαν αυτές τις δυνατότητες. Νομολογία και το πόσο ε, αυξάνεται ο όγκος αυτής. Ναι, πρέπει να δώσουμε ε, κάποιες κατευθύνσεις στους νομικούς και να συνεργαστούμε με τη Eurojust για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε συνόψεις της νομολογίας και να έχουμε και μια κοινή μεθοδολογία εργασίας για να αξιολογούμε τις συνθήκες κράτησης. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουν από τη βάση δεδομένων οι επαγγελματίες. Αυτά. Ο κύριος Βηγιαρέχου. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα σας ε, δώσω μία γενική σφής απάντηση από πρακτική σκοπιά. Οι υποθέσεις που μας απασχολούν, περίπου 600 υποθέσεις πέρσι, είναι διμερείς υποθέσεις οι περισσότερες ε, τουλάχιστον. Διευκολύνουμε βεβαίως την εκτέλεση άλλων ενταλμάτων σύλληψης, δηλαδή στην προηγούμενη Τρίτη είχαμε μία Action Day και ε, χρειάστηκε να εκδοθούν έξι επιπρόσθετα εντάλματα σύλληψης επιτόπου σε σχέση με τον αρχικό αριθμό που ήταν προγραμματισμένος. Έχουμε να κάνουμε με διαφορετικά σενάρια. Αυτό είναι το απλούστερο που σας αναφέρω. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε με τις ε, πιο ε, επίγουσες περιπτώσεις και βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εκτέλεση, η εκτέλεση της ε, απόφασης σε πολλές περιπτώσεις βεβαίως δεν υπάρχει συμμόρφωση. Υπάρχει η απόφαση η οποία έχει επικαιροποιηθεί, αλλά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συμπληρώνει αυτό το νομικό πλαίσιο. Η περίπτωση Αρανιώσα Καλταράρο ε, οδήγησε σε ερμηνεία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η απόφαση Πετρούχεν μας ε, έθεσε άλλες προαπαιτήσεις για ε, περιπτώσεις, για αιτήσει έκδοσης όταν ο πολίτης προέρχεται από μία τρίτη χώρα. Αλλά οι αρχές μας, οι δικαστικές μας αρχές χρειάζονται την υποστήριξή μας γιατί είναι δικαστές και εισαγγελείς αλλά πρέπει να έχουν μία εις βάθος γνώση της νομολογίας του Δικαστηρίου του Λουξεμβούρου και ε, επίσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούρου γιατί στην περίπτωση Ρομέρο και η απόφαση Χαουλεγγύ ήταν πολύ προσήκουσες και πρέπει να έχουμε πίκερες πληροφορίες, ε, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό ε, η Eurojust μπορεί να συνδράμει. Χρειαζόμαστε προδιαγραφές σε σχέση με την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα, τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές. Και κάποια στιγμή χρειάστηκε να αξιολογήσουμε και την ανεξαρτησία της εισαγγελική αρχής. Και το Συμβούλιο της ε, Ευρώπης εκδίδει ε, αποφάσεις και εκθέσεις, αλλά θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να συνδράμει και η Eurojust με βάση την ε, πιο πρόσφατη νομολογία και με βάση την τελευταία απόφαση για τις δικαστικές αρχές της 12 Δεκεμβρίου είναι μια πολύ σαφής απόφαση σε σχέση με το πώς ο εισαγγελέα μπορεί να εκδώσει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη νομολογία γιατί αυτό μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς λειτουργεί αμοιβαία αναγνώριση. Χρειαζόσαστε εισαγγελείς. Είναι το, το λάδι που κάνει τη μηχανή να λειτουργήσει οι εισαγγελικές αρχές. Δηλαδή, ο εισαγγελέα προωθεί κατά δυναμικό τρόπο την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων. Και αυτό σε πλήρη συμμόρφωση των οδηγιών και τη διπλή εκπροσώπηση της, που προβλέπεται από την οδηγία του 2010 που έχει εφαρμοστεί στα περισσότερα κράτη-μέλη και λειτουργεί πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βιαρέχο και σας ευχαριστούμε όλους. Ε, ζητούμε συγγνώμη για το, την πίεση χρόνου, αλλά έχουμε υπερβεί και το χρόνο μας. Προβλεπόταν ε, ε, μέχρι τις 10.30 γιατί είσαστε εδώ για να ανταποκριθείτε στα θέματα και ανησυχίες μας, διότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ασχολείται εις βάθος με αυτό το θέμα της εκτέλεσης ε, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Άρα η παρουσία σας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Δυστυχώς έχουμε υπερβάσει συνέχεια στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ο κύριος ε, Θαρθαλέχος έχει το λόγο για, τις, ε, για τα καταληκτικά σχόλια. Σημερίζομαι τα σχόλια των εισηγητών τη στιγμή που μιλάμε για πληροφορίες, πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή του πλαισίου, φυσικά μας ενδιαφέρει η, η εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ότι αυτό το μέσο δικαστικής συνεργασίας είναι μια μεγάλη επιτυχία και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πολύτιμο μέσο με σύνεση και να το βελτιώσουμε. Και Γι' αυτό ακριβώς μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε τους τομείς όπου θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Βεβαίως, τα προβλήματα που ε, θέτει η απόφαση πλαίσιο είναι ακριβώς αυτής της φύσης όπως το θέμα της μεταφοράς στην Εθνική Ενωμητάξη. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε λόγος για το διπλό αξιόπινο το οποίο είναι ένα ε, θέμα το οποίο στρέβλωσε την ε, εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης το θέμα της αναλογικότητας που κατά περίεργο τρόπο δεν αναφέρεται στην απόφαση πλαίσιο, αλλά που είναι ύψης της σημασίας και που πρέπει να μας απασχολήσει στα πλαίσια ανάπτυξης άλλων μέσων δικαστικής συνεργασίας έγινε λόγος για το γλωσσικό καθεστώς, την προετοιμασία των δικαστών, την διαδικασία διαβούλευσης και ο κύριος ε, Χιμένεφ Βιαρέχο μίλησε και για το ρόλο της Eurojust στα πλαίσια αυτά. Όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα στοιχεία για να προχωρήσουμε με την εργασία μας και είναι μία εργασία στο ύψος των περιστάσεων και της εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και φυσικά το θέμα της εμπιστοσύνης είναι ύψη σημασία στην ε, συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πολύ συνεπτικός και βεβαίως ευχαριστούμε τους τρεις πανελίστες. Σίγουρα το σημείο αυτό είναι μια κρίσιμη παντή ε, για την περαιτέρω δουλειά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για το θέμα αυτό που χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ μας για θέματα κανόνων και προτύπων. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η κοινή συνάντηση με την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ και την Επιτροπή Ντρουά για την αποστολή που πήγε ε, στο φόρουμ ε, για τους πρόσφυγες στη Γενέβη. Σε ένα λεπτό.